Day, and then I'll move in, into NOC. Dear colleagues, good afternoon. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Προτείνω να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ε, το σημείο 2 της ημερησίας διατάξεως, το οποίο ε, αφορά τις εκθέσεις που και την ε, αναφορά για την Ίσπρα, μάλλον το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως, να το κάνουμε κάποια άλλη φορά, έτσι ώστε να το συνδυάσουμε με τις επισκέψεις στο Λουξεμβούργο και, στο, και στην Γαλλία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή ανταλλαγή γενική πληροφοριών και απόψεων. Αντιτίθεται κανείς, όχι. Να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε 16 ε, ε, γλώσσες και είναι web streamed η συνεδρίασή μας. Επίσης, να σας πω ότι τα πρακτικά της 5ης Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας και ε, μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει σχόλια. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γκρούντλερ από το Μίσιγκαν και την Ουάσιγκτον ο οποίος ε, εκπροσωπεί την ΕΙΠΑ, η οποία είναι ε, η ε, οργάνωση για το περιβάλλον. Μέχρι πέρσι δεν ξέραμε και πολλά πράγματα για αυτήν ε, την υπηρεσία, αλλά τώρα νομίζω ότι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι ένα Ινστιτούτο ε, το οποίο είναι γνωστό, το οποίο επηρεάζει. Ε, θα σας δώσω το λόγο λοιπόν έτσι ώστε να κάνετε μια πρώτη γενική παρέμβαση και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου για την ε, για οποιαδήποτε που, που ελέγχει συγγνώμη το, την εκπομπή ε, ρήπων από ε, ε, οποιοδήποτε μέσο και επίσης ε, κυρίως ασχολούμαστε με τα σωματίδια και τους ρήπους που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα, από τα ε, μικρά και μεγάλα φορτηγά, από ε, φορτηγά, από ε, τρακτέρια, άλλα αγροτικά μηχανήματα κτλ. Οτιδήποτε δηλαδή κινείται και προκαλεί, παράγει μόλυνση, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Ε, μας ενδιαφέρει επίσης ε, να βρούμε λύσεις, ε, να κάνουμε μετρήσεις και να υποστηρίζουμε οποιασδήποτε λύσεις. Καθορίζουμε τα, τα όρια, τα αποδεκτά όσον αφορά εκπομπές αερίων από οποιοδήποτε μηχάνημα, από αέρος και χερσαίο καθορίζουμε στρατηγικές και επίσης ελέγχουμε μέσω ε, έρευνας ε, τις ενδεχόμενες εξελίξεις. Το κύριο εργαστήριό μας βρίσκεται στο Μίσιγκαν και υποστηρίζει ε, όλες τις προσπάθειές μας καθώς και τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε. Ε, είναι μεγάλη η τιμή μου ε, που έχω την δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με έναν ε, ιστορικό φορέα και που έχουμε ήδη συνεργαστεί σε κάποια συγκεκριμένα ε, προγράμματα τα οποία έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ ε, καλά. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα ε, η EPA βάσει της νομοθεσίας για τον καθαρό αέρα έχουμε ξεκινήσει διάφορες τεχνολογικές διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν τις τεχνολογικές απαιτήσει, ε, κυρίως όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, μάθαμε ότι τα στάνταρ τα οποία βασίζονται στις επιδόσεις ε, μαζί με κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά σχεδιασμού μπορούν να δώσουν και καινοτομία αλλά και καλή τεχνολογία. Το δεύτερο που μάθαμε είναι ότι ο καθορισμός των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 ο καθορισμός αρχών που θα διέπουν και την κατασκευή των αυτοκινήτων αλλά και την ποιότητα των καυσίμων ε, ε, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ε, έχουμε επίσης ασχοληθεί με την, τον έλεγχο των επιδόσεων των καυσίμων. Τρίτον, κάνουμε ένα μοντέλο παρακολούθησης των τεχνικών διεργασιών έτσι ώστε ε, να υπάρχει διαφάνεια. Μας ενδιαφέρει ε, να ε, είναι, να μας ενδιαφέρει οι Αμερικανοί πολίτες να ευνοούνται από τις ε, αποφάσεις που παίρνουμε. Θεωρούμε ότι είναι δικιά μας υποχρέωση να υλοποιούμε με πολύ σοβαρό τρόπο οτιδήποτε αναφέρεται στην, στους κανονισμούς και την νομοθεσία για τον καθαρό αέρα. Και αυτό το κάνουμε γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει καθαρός αέρας για τους πολίτες δεύτερον, ε, γιατί εάν αυτό δεν λειτουργήσει, σημαίνει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερε προσπάθειε, ε, πράγμα που ενδεχομένω θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και οπωσδήποτε θα προκαλέσει ε, διαδικασίε χρονοβόρε και ακριβέ τα προγράμματά μας για τα αυτοκίνητα αλλά και για τα φορτηγά λειτουργούν μέχρι τώρα. Γνωρίζουμε ότι ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς την ποιότητα, αλλά παρόλα αυτά εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πάρα πολύ βελτιώσει τις επιδόσεις μας βάσει ακριβώς των αποτελεσμάτων που έχουν δώσει τα προηγούμενα χρόνια τα προγράμματά μας. Ε, ε, μαθαίνουμε μαθήματα από το παρελθόν, κάνουμε νέες τεχνολογικές εξελίξεις κλπ. Ε, τι έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει ότι ε, είναι, σημαντικά, τα, είναι σημαντικές οι δοκιμές. Ε, στη δεκαετία του 90 η EPA έφτασε, έβαλε κάποιες διαδικασίες ακόμα και ενώπιον των δικαστηρίων έτσι κυρίως για ελαφρά οχήματα αλλά ακόμα και για βαρέα οχήματα. Το 1995, το 1998 αλλά και το 1999 η οι που είχαμε και οι διαδικασίες που είχαμε ε, αναλάβει οδήγησαν σε κάποιες ε, συμφωνίες ε, οι οποίε οδήγησαν σε μια καλύτερη νομοθεσία για τον καθαρό αέρα και πληρώθηκαν κάποιες κυρώσει οι οποίες ήταν πάρα πολύ υψηλές. Επίσης η EPA μετά δημιούργησε μια, κάποιες νέες διαδικασίες δοκιμασιών για τα ελευθερά αλλά και για τα βαρέα οχήματα ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και κάποιες διαδικασίες οι οποίες αφορούσαν τον, τον καλό τρόπο οδήγησης. Η EPA επίσης αύξησε ε, όλες τις διαδικασίες ε, ε, ελέγχου και αδειοδότησης όσον αφορά και τα βαρέα αλλά και τα ελαφρά οχήματα. Ένα άλλο αποτέλεσμα που είχαμε ήταν ότι πολλές εταιρείες και για ελαφρά αλλά και για βαρέα οχήματα ξεκίνησαν και υιοθέτησαν εσωτερικές διαδικασίες ε, έτσι ώστε να καλύψουν ενδεχόμενα προβλήματα η EPA ε, ε, ε, καθόρισε, κάποια στάνταρ όσον αφορά την, το, τη διάρκεια ζωής των αυτοκινήτων από 120.000 μέχρι 150.000 μίλια για τα αυτοκίνητα. Αυτά τα στάνταρ έχουν υπολογιστεί με βάση όλα τα στοιχεία των οχημάτων και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το αμερικανικό πρόγραμμα είναι ισχυρό γιατί ακριβώς βασίζεται ε, σε, μεγάλο βαθμό ε, στην ε, νομοθεσία για τον καθαρό αέρα και δίνει στην EPA συγκεκριμένες δυνατότητες ελέγχου των αυτοκινήτων, των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ξεκινούν ε, τα τεστ, οι δοκιμές αυτές ε, πριν ε, από την παραγωγή, στη διάρκεια της παραγωγής μέχρι το τέλος της παραγωγής τους. Ε, επίσης ε, ε, έχουμε συγκεκριμένες δοκιμασίες, τεστ που αφορούν πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Επίσης μετά από ενός έτους χρήση και μετά από τέσσερα έτη χρήσης του αυτοκινήτου πρέπει να περνούν ξανά από συγκεκριμένα τεστ και δοκιμές. Ε, πρόσφατα αφού καθορίστηκαν από την EPA ε, κάποια πρώτα πρότυπα όσον αφορά τις, ε, τα αέρια του θερμοκηπίου προχωρήσαμε έτσι ώστε να καλύψουμε και τη, τους ρήπους εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Αυτά, αυτές οι δοκιμές είχαν σαν αποτέλεσμα ότι κάποιες εταιρείες και αμερικανικές αλλά και διεθνείς είχαν δώσει κάποια στοιχεία όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμων ή όσον αφορά ε, τις επιδόσεις οι οποίες δεν ήταν σωστές. Ε, Από τη στιγμή που ε, μάθαμε πλέον το μάθημα με την περίπτωση της Volkswagen, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη και τρόπους και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούν να προβλέψουν οι κατασκευαστές. Πέρσι διευρύναμε ε, το, ε, το ε, έτσι ώστε να βάλουμε και κάποια νέα τεστ, κάποιες νέες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη ακριβώς τις διαφορετικές τεχνολογίες, τις εξελίξεις κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης η επιβολή του νόμου. Δηλαδή μπορεί κανείς να έχει πάρα πολύ αυστηρά στάνταρ όσον αφορά τις εκπομπές μπορεί να έχει πολύ αυστηρά τεστ και δοκιμές κτλ. Αλλά όλα αυτά ε, δεν ε, μπορεί να έχουν κανένα αποτέλεσμα εάν ε, δεν επιβάλλεται με κάποιο τρόπο η χρήση τους και τα καλά τους αποτελέσματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να λειτουργήσουν από κοινού γιατί διαφορετικά με μονομένα στοιχεία δεν μπορεί να δώσουν αποτέλεσμα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να έχει κανείς τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις, ε, δηλαδή ε, η ουσία των προτύπων ανάπτυξης και συμμόρφωσης τα οποία εμείς έχουμε αναπτύξει, καθώς επίσης και όλη αυτή η εργασία η οποία σχετίζεται με τις δοκιμές βασίζεται σε μια τεχνογνωσία την οποία έχουμε αναπτύξει, σε προσωπικό το οποίο είναι γνώστες. Επίσης έχουμε δημιουργήσει δημιουργήσει ένα εργαστήριο το οποίο λέγεται National Vehicle and Fuel Emissions Laboratory ε, στο Michigan, στην περιοχή Ann Arbor. Ε, έχουμε ε, προσωπικό το οποίο είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένο και τεχνικά εξοπλισμένο έτσι ώστε να κάνει αυτού του είδους ε, τις ε, ε, μελέτες και δοκιμές. Το σημαντικό για μας είναι να κρατήσουμε, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στο κοινό όσον αφορά τον καθαρότερο αέρα. Πρέπει να σας πω ότι συχνά εμείς αναφερόμαστε στην προσέγγιση μας ως ένα σχήμα 3x3. Δηλαδή, το πρώτο 3 αναφέρεται στις δοκιμές που κάνουμε και που μπορούν να, να οδηγήσει, μπορεί να οδηγήσει σε ε, δοκιμές σε τρία σημεία ε, της, ε, του κύκλου ζωής της, του, του οχήματος. Δηλαδή, όσον αφορά, ο πρώτος έλεγχος θα αφορά τα πρωτότυπα, ο δεύτερος έλεγχος θα αφορά τα καινούργια οχήματα και το, ο τρίτος έλεγχος θα αφορά τον έλεγχο του οχήματος αφού θα έχει κυκλοφορήσει στον δρόμο για κάποια χρόνια. Επίσης, ε, ε, ε, το επόμενο τρία αναφέρεται στους τρεις διαφορετικούς τύπους δοκιμών που κάνουμε. Πρώτον, όσον αφορά τις εκπομπές, δηλαδή βάση των δοκιμών δυναμομέτρου. Δεύτερον, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο στο δρόμο. Και τρίτον, είναι κάποια περίεργες, κάποιες περίεργες δοκιμές, τις οποίες, ε, και τις οποίες δεν ε, ε, γνωστοποιούμε στους κατασκευαστές. Εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι στην 40χρονη ιστορία του προγράμματός μας διαρκώς ενημερώνουμε και επικαιροποιούμε την προσέγγιση μας όσον αφορά αυτές τις δοκιμές και τις συμμορφώσεις. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό και ότι αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ευελπιστώ σε μια καλή ανταλλαγή ε, απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε σκεφτόμαστε στην Ευρώπη ότι έχουμε τους καλύτερους περιβαλλοντικούς νόμους, καλύτερους νόμους για τους καταναλωτές, αλλά ακούγοντα τη δική σας ε, παρέμβαση έχουμε πολλά να μάθουμε από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε στους τομείς αυτούς. Να περάσω τώρα ε, στα μέλη της Επιτροπής. Ε, δυστυχώς ο ένας εισηγητής ε, λείπει σε αποστολή και ο κύριος Άλβα ο δεύτερος εισηγητής, έχει κολλήσει σε ένα μποτιλιάρισμα. Θα του δώσω το λόγο όταν έρθει. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Κρόνβλερ, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γερμανικά, αλλά θα σας μιλήσω στα γερμανικά, γι' αυτό αν θέλετε να βάλετε τα ακουστικά σας. Έχουμε και διερμηνία. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα και χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ. Ο εισηγητή μα δυστυχώ έχει μείνει στην κίνηση, έχει κολλήσει. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά θα έρθει, οπωσδήποτε θα έρθει. Αυτό που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι είπατε. Ε, στην Ευρώπη θα έχουμε διαφορετική νομοθεσία και αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ακριβώ ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ Αμερικανική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλο τη δική σα υπηρεσία, πείτε μα σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ε, προτύπων για το περιβάλλον και των συγκεκριμένων <coughs> στόχων για την ατμόσφαιρα. Ποια είναι η δική σας λοιπόν η αρμοδιότητα και το δικό σας καθήκον ως υπηρεσία. Η e η EPA ασχολείται και με την ε, ατμόσφαιρα, δηλαδή πόσο καθαρός πρέπει να είναι ο αέρας και τις σχετικές προδιαγραφές, όπως επίσης και με νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών, προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς, ε, τη συγκέντρωση των ρήπων στην, στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η δική μου συγκεκριμένη ευθύνη ε, είναι ο καθορισμός αυτό της νομοθεσίας για τις κινητές πηγές, δηλαδή για τα επιβατικά οχήματα και άλλου είδους ε, μεταφορές που είναι πηγές ε, ρήπων για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά αυτούς τους στόχους ε, της βελτίωσης του ατμοσφαιρικού αέρα στις διάφορες, σε διάφορα μέρη της ε, αμερικανικής επικράτειας. Επίσης, ε, το θέμα του εξοπλισμού και από εκεί προέρχονται ε, διάφοροι ρήποι. Προσπαθούμε επίσης σε ζητήματα πιστοποίησης να, υπάρξει, να υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης όταν υπάρχουν προβλήματα να διερευνώνται και να προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει παραβίαση νομοθεσίας. Η EPA λοιπόν έχει πολύ ευρία αρμοδιότητα υπό την αμερικανική νομοθεσία όχι μόνο για να ορίζει το, το, για να το πόσο καθαρός πρέπει να είναι ο αέρας για την ανθρώπινη υγεία, αλλά ε, και ποιες είναι οι βασικές πηγές της ατμοσφαιρικής αυτής ρήπανσης. Ναι, αλλά είσαστε υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο. Δεν είσαστε ερετό ε, εκλεγμένο. Ε, σε εμά τα πρότυπα αυτά καθορίζονται με έγκριση του Κοινοβουλίου. Πού βρίσκεται λοιπόν στη δική σας περίπτωση, στα ό,τι τη χάραξη των οριακών τιμών, ε, η δημοκρατική νομιμοποίηση, πώς ε, το διασφαλίζεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Το Κογκρέσιο ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, το 1970 ε, ψήφισε τον, την νομοθεσία για τον καθαρό αέρα και δίνει το καθήκον στην EPA να διεκπεραιώνει τις αρμοδιότητές της. Βάσει αυτής της νομοθεσίας λοιπόν και έδωσε, τη δυνατό, έδωσε σε εμά το καθήκον να ορίσουμε αυτές τις προδιαγραφές και να τις εφαρμόσουμε. Η κυβέρνηση έχει εκχωρήσει κάποιες ε, αρμοδιότητες ε, στο δικό μου επίπεδο για να μπορέσω και να ορίζω αλλά και να επιβλέπω την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν οριστεί οι οριακέ τιμέ. Δεν αναμειγνύονται πλέον στην όλη διαδικασία οι βουλευτέ τα πρότυπα αυτά ορίζονται από εσά, από την EPA, από την υπηρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ συναρπαστικό το γεγονό ότι ε, περιγράφεται ότι συμμετέχει και η δημόσια, η κοινή γνώμη. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη μέσω τη διαδικασία διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ συμμετέχει λοιπόν η κοινή γνώμη στη δική σα περίπτωση, και δεύτερη ερώτηση, σε τι βαθμό συμμετέχει και ο βιομηχανικό κλάδο σε ό,τι αφορά τον ορισμό των οριακών τιμών, γιατί είπατε στην τελική ανάλυση performance based. Θα πρέπει δηλαδή δηλαδή να είναι δυνατόν στην πράξη να τηρούνται οι ουριακέ τομέ ε, που ορίζονται. Καταρχά, λοιπόν, πείτε μου ε, πώς συμμετέχει η κοινή γνώμη και πώς συμμετέχει και ο βιομηχανικό κλάδος. um, Προφανώς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό επίβλεψη ε, ομοσπονδιακών ε, ε, υπηρεσιών σαν τη δική μα, την EPA, και προφανώς γίνονται ακροάσεις σαν αυτή, κάνουν ερωτήσεις στου υπαλλήλου της EPA πώ ορίζουν αυτές τι προδιαγραφέ. και έτσι έχουμε αυτή την εξουσία. Τώρα το πώς ε, την ασκούμε αυτή την εξουσία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μια πολύ ανοιχτή και διαφανή διαδικασία με δημόσιε συνεδριάσεις αλλά και πριν από την πρόταση για μία προδιαγραφή. Ε, κατά την ανάπτυξη αυτή τη προδιαγραφή έχουμε μία πολύ συνεργατική διαδικασία. Από ε, με μη κυβερνητικέ οργανώσει, με βιομηχάνους, με ε, ολόκληρη την ε, αλυσίδα ε, διανομή, όπω επίση και με την κυβέρνηση. Γιατί πιστεύουμε ότι μία τέτοιου είδου συνεργατική και διαφανή προσέγγιση θα ενημερώνει καλύτερα του υπεύθυνου λήψη αποφάσεων. Οπότε έχουμε τι συζητήσει, δημόσιε συζητήσει συζητήσεις, δημόσια κροάσεις, ε, ε, ε, λαμβάνουμε σχόλια και γραπτά και προφορικά και έχουμε μία υποκρέωση να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα σχόλια και να τους εξηγήσουμε πώς τα λάβαμε υπόψη όταν λάβαμε τις τελικές μας αποφάσεις. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις απαντήσεις που μας δώσατε, αλλά και για την παρουσίασή σας. Στην ερώτηση 10, στην απάντησή σας είπατε ε, είπατε ότι το ευρωπαϊκό τεστ EDC είναι μη επαρκές ε, για την ε, για, για την, την ανείχνευση των εκπομπών ήδη θεωρούσατε ότι είναι παροχημένο από τη δεκαετία του 90. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι τόσο παροχημένες και ανεπαρκείς αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούμε επειδή δεν καλύπτει επιθετική οδήγηση σε μεγάλες ταχύτητες ή γιατί θεωρείτε ότι δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της ε, ε, οδικής συμπεριφοράς του ε, αυτοκινήτου ο έλεγχος. Ναι, είναι η απάντηση. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ απαιτητική αυτή η διαδικασία όσον αφορά στο όχημα γιατί ο βαθμός επιτάχυνσης, ε, η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, η ε, έλλειψη της ε, χρήσης του κλιματισμού. Έχουμε πέντε κύκλους δοκιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους χρησιμοποιούν στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο, σε κρύες θερμοκρασίες, σε υψηλές θερμοκρασίες με τον κλιματισμό αναμένο και οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, επιθετική οδήγηση. Αυτές είναι κανονικές συνθήκες λειτουργίας του ε, αυτοκινήτου και η ιδέα μεταξύ αυτών των πέντε κύκλων δοκιμών είναι να, να ε, βασίσουμε σε αυτές το σχεδιασμό των, των αυτοκινήτων Όταν Αν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα έπρεπε να επιτύχει κάποιους στόχους σε αυτές τις πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, προσπαθούμε να το επιτύχουμε όταν όλοι οι καταναλωτές ε, χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. και σήμερα αναφερθήκατε ε, στην ε, τεχνολογική εξέλιξη. Υπάρχουν στοιχεία στο παρελθόν που κατέστη σε ακόμη πιο ανεπαρκή και παροχημένους, ε, ανεπαρκής και παροχημένους ελέγχους. Ε, το NDC e και ε, το, ο κύκλος ε, ε δυναμομετρικής πέδησης ήταν κάτι το οποίο ήδη από την αρχή της λειτουργίας αυτές οι διατάξεις δεν μπορούσαν να δεχθούν ένα επίπεδο ε, επιτάχυνσης. Υπήρχαν, ε, ήταν λοιπόν δοκιμές που ε, ήταν διαφορετικές από τα σύγχρονα δυναμόμετρα που μπορούν την επιτάχυνση, την επιβράδυνση να τη χειριστούν πολύ καλύτερα ενώ αρχικά ε, ήμασταν βασισμένοι ε, στο τι μπορούσε ο εξοπλισμός να αντέξει και όχι το όχημα. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να υπάρχουν επιπλέον ε, οχήμα, δοκιμές στα οχήματα. Κάτι επίσης που διαπιστώσαμε από την εμπειρία μας από την αρχή ήδη με τις διατάξεις αναστολής είναι κακή ερμηνεία ότι έπρεπε να επιτύχουν απλώς ε, τις, ε, τους στόχους ε, των εκπομπών σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, γιατί αυτό αναφερόταν στη δοκιμή και διαφωνούμε εμείς με αυτή την ερμηνεία και εμείς στις διαδικασίες επιβολής μας θελήσαμε να υπάρξουν επιπρόσθετοι κύκλοι δοκιμών για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα και συγκρούσεις. Στη γραπτή σας απάντηση αναφερθήκατε επίσης και στο πρόγραμμα επίβλεψης των Ηνωμένων Πολιτειών ε, με μη συμβατικές ε, μεθόδους ελέγχου και ε, στην κίνηση του αυτοκινήτου στον δρόμο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Πώς μπορείτε να το συνδυάσετε αυτό με τη διαδικασία της συνήθεια έγκρισης τύπου. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Ευχαριστώ. Εμείς δεν θέλουμε οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ε, να ξέρουν ε, όλα τα μυστικά ε, των, κύκλων δοκιμών μας. Γι' αυτό ακριβώς τα αναμειγνύουμε, τα αλλάζουμε, ε, προσπαθούμε να σκίσουμε ένα όχημα με διαφορετικούς τρόπους, να το δούμε με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς τρόπους, ε, με όσους μπορούμε να σκεφτούμε, να είμαστε απρόβλεπτοι. Είμαστε η νέα απρόβλεπτη EPA και αποκαλούμε τους εαυτούς μας έτσι για κάποιο λόγο. Ε, κατά τη δική μας άποψη, οι εκπομπές που αναπνέει ο κόσμος πρέπει να μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές που προκύπτουν από τον εργαστηριακό έλεγχο. Αυτή είναι η βάση της προσέγγισης μας και αν όχι τότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ε, είτε το εργαστηριακή μέθοδος είναι προβληματική είτε το όχημα. Σε κάθε περίπτωση εγώ ε, θα ήθελα να είμαστε περίεργοι ως προς αυτό, να ενδιαφερθούμε, να διερευνήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και αν υπάρχουν ζητήματα να τα αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Σχάλτε Μόζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω α, τον κύριο Γκρούντλερ που έχει φτάσει, που έχει έρθει εδώ πέρα και νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμε οι εμπειρίε που μα ε, δίνετε δίνεται για να βελτιώσουμε και την ειδική μα ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολλά θεωρώ ότι μπορούμε να μάθουμε από εσά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα τι γραπτέ σα απαντήσει και μετά από με αυτά που μα είπατε κιόλα. είναι ότι δεν θέλετε η παραγωγή οι βιομήχανοι να ξέρετε ακριβώς το πώς γίνονται οι έλεγχοι για να μην υπάρχει δυνατότητα να τους ε, υπονομεύσουν. Από πότε έχετε αναπτύξει τέτοιου είδους ε, νοοτροπία, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η ατμόσφαιρα υποψία και καχυποψίας κατά των βιομηχάνων και των κατασκευαστών. Για πείτε μας λίγο κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα ελέγχου δοκιμών και κατά το παρελθόν και σήμερα είναι στοχευμένο. Και αυτό που έχουμε μάθει από την εμπειρία αυτή τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο πρόβλεπτοι. Να έχουμε ένα τέτοιο στοιχείο μη προβλεψιμότητα. Γιατί δεν υπήρχαν αυτοί οι κινητήρες το 2009. Τότε που ξεκίνησαν, κάναμε πάρα πολύ σχολαστικού σχολαστικούς ελέγχους. Αν είχαμε τότε κάνει έλεγχο και με τους συσκευές PIMS, θα έχουμε σίγουρα ανακαλύψει αυτές τις συσκευές ε, παράκαμψης. το κάναμε όμω ε, μόνο για τα φορτηγά, γιατί από, τότε, από εκεί προέρχονται οι πιο πολλέ εκπομπέ ε, ρήπων ε, στην Αμερική. Άρα, στάσαμε προτεραιότητε τότε και λάβαμε αποφάσει και μάθαμε από τα παθήματα του παρελθόντο. Και στείλαμε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μια επιστολή σε όλου του κατασκευαστέ αυτοκινήτων ότι πρόκειται να υιοθετήσουμε νέες ε, διαδικασίες δοκιμών και θα κρατούσαμε τα οχήματά τους λίγο παραπάνω και δεν ε, τους εξηγήσαμε γιατί. Έτσι λοιπόν ε, προσεγγίζουμε το θέμα των ελέγχων και πριν και μετά την κατασκευή. Τώρα πλέον λοιπόν ακολουθούμε αυτή τη διαφορετική προσέγγιση. Κοιτάξτε, η ερώτηση κ. Σαλντεμόζε. Πιστεύετε ότι είναι στη φύση του κατασκευαστή του αυτοκινητοπαραγωγού να τηρεί μόνο το, τα ελάχιστα πρότυπα, το λιγότερο που είναι δυνατόν. Γιατί είσαι τόσο καχύπτωπο δηλαδή. Στα τέλη δεκαετία του 90 η απάντηση. Χρησιμοποίησαμε τις τεχνικές για να καταπολεμήσουμε αυτές τις συσκευές υπονόμευσης και νομίζω ότι ε, το έμαθαν το μάθημα γιατί ήταν πάρα πολύ ε, οδυνηρό από οικονομικής άποψης να μην τηρούν τις προδιαγραφές. Όταν καταλήγουν δηλαδή τα πρόστιμα να είναι σε ύψη δισεκατομμυρίων για ομίλους, ε, πλέον είναι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το στοιχείο αυτό. Και άρα δεν πιστεύω ότι είναι στη φύση του να κάνουν αυτό, να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Και κοιτάξτε, να σα πω ότι σε σχέση με τη δεκαετία του 90, μια εταιρεία μου είπε ότι υπήρχε και μια ειδική επιτροπή ε, για τις συσκευές αυτές παράκαμψης ε, σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία κατασκευής. Άλλες εταιρείε προβάλλουν το τι ακριβώς εννοείται με τις συσκευές αυτές. Φέτος εμείς λοιπόν ζητούμε από κάθε εταιρεία να έρχεται να μας ενημερώσει τι δικασία ακολουθείτε για να αποφευχθούν τέτοιες συσκευές. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για τις συσκευές, για τον έλεγχο των εκπομπών που θα χρησιμοποιήσουμε. Εσείς όμως έχετε όλες αυτές τις διαδικασίε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπορία, τη διάθεση στο εμπόριο θα συστήνετε λοιπόν και στην Ευρώπη τέτοιου εκτενεί ελέγχου και δοκιμέ. Κοιτάξτε, είμαι μηχανικό και οι μηχανικοί φυσικά πάντα θέλουν όλο και πιο πολλά δεδομένα. Και όπω είπατε, στην Αμερική είμαστε αρκετά αδιάκριτοι. Γι' αυτό έχουμε όλε αυτέ ε, τι δοκιμέ σε όλα αυτά τα επίπεδα. Εγώ τώρα πώ να σα πω τι να κάνετε. Εγώ είμαι Αμερικάνο. Πώ θα βγω να πω στου άλλου τι να κάνουν. Και δεν είμαι ειδικό για τι δικές σας προτάσεις. Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας πω ότι και σε ό,τι αφορά το RDE και σε ό,τι αφορά τη δικασία ελέγχου και δοκιμών τύπου είναι σωστή η κατεύθυνση που ακολουθείτε. Οι πιο πολλέ δοκιμέ είναι η σωστή προσέγγιση, ιδιαίτερα σε περίπτωση γι' αυτή. Έχουμε μια εταιρική σχέση και με τους συναδέλφους από την Καλιφόρνια και από τον Καναδά για να υπάρχει καλύτερη υποπτία τη όλη διαδικασία για να ξέρουμε ποιος ελέγχει τι και να γίνεται ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μάκερ. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Γκρούντερ. Ναι, μιλάω Ολλανδικά. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Είναι σαφέ ε, ότι το αμερικανικό σύστημα διαφέρει σε αρκετά σημεία από το ευρωπαϊκό. Και αυτό που είναι σημαντικό, πιστεύω, είναι να ξέρουμε γιατί έχουν γίνει συγκεκριμένε επιλογέ, με, ποια, με ποια επιχειρηματολογία. Να το κατανοήσουμε λοιπόν αυτό για να μπορέσουμε να εξαγαγούμε τα απαραίτητα συμπεράσματα και πορίσματα. Θα ήθελα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό να θέσω τα εξή ερωτήματα. Οι ακροάσεις εδώ κατέδειξαν με σαφήνεια ότι σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τον έλεγχο των εκπομπών, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους είναι η μείωση του διεξοδίου του άνθρακα. Των εκπομπών διεξοδίου του Και αυτό φαίνεται ότι είναι ε, μια βασική ε, διαφορά με την Αμερική, όπου εξ αρχής η μείωση των όξι ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Πείτε μας λοιπόν πώς ε, αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό των ε, αζωτούχων σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρτίζουμε λοιπόν και ε, ορίζουμε τα όρια και τα πρότυπα για τις εκπομπές και των νόξ και των διοξιδίων του άνθρακα και βάσει τεχνικών στοιχείων. Κάνουμε τεχνικές μελέτες, κάνουμε ε, μοντέλα προσωμείωσης οχημάτων, κάνουμε μελέτες ε, οικονομικού αντικτύπου και αναπτύσσουμε λοιπόν πρότυπα βάση απόδοσης, δηλαδή τι ε, πρότυπα χρειάζεται να ακολουθούνται προκειμένου να τηρούνται τα όρια νοξ και διοξιδίου του άνθρακα βάσει τη σχετική νομοθεσία για την ε, ρήπανση τη ατμόσφαιρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ διαφανή αυτή η δικασία για τον καθορισμό των προτύπων αυτών. Έχουμε ακούσει τώρα στο παρελθόν διάφορα ε, επιχειρήματα ότι το, η υπηρεσία μα, η υπηρεσία προστασία του περιβάλλοντο, θα πρέπει να επιλέξει είτε μείωση του NOx είτε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, κοιτάξτε, ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία εμείς τα απορρίπτουμε τα επιχειρήματα αυτά. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η τεχνολογία για να μειωθεί και η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και τον Όξο εκ παραλλήλου. Και αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε. Ο κ. Τεμέης Μάκρης, μάλιστα, είναι λοιπόν διαφορετική προσέγγιση σας. Συμφωνείτε όμως με την ανάλυση την εξή ότι Ανάλογα με το πώ ορίζονται τα πρότυπα για τι εκπομπές NOx ή διοξιδίου του άνθρακα, ε, προσαρμόζουν και η αυτοκινητοπαραγωγή τη διαδικασία παραγωγής αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα, τα δίζελ και τα μετσινοκίνητα. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι μάλλον διαφωνώ με αυτό, με τον όλο το σεβασμό που σας τρέφω έχουμε ορίσει τα όρια και για τα ζωτούχα και για το διοξείδιο του άνθρακα, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Κάνουμε τη δουλειά μα για να φροντίσουμε να είναι εφικτά φυσικά τα όρια αυτά. Αλλά μετά επαφείται στον ε, αυτοκίνητο παραγωγό να επιλέξει την προηγμένη τεχνολογία, για παράδειγμα βενζίνη, δίζελ, ε, υβριδικά. Όλα αυτά επιτρέπονται λοιπόν στις ΗΠΑ για να επιτευχθούν τα πρότυπα που έχουν τεθεί, δεν ε, προτιμούμε τη μία ή την άλλη τεχνολογία. Και να σας υπενθυμίσω ότι τα αυτοκίνητα ε, diesel έχουν την ίδια απόδοση με τα ε, μετζινοκίνητα σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ. Εμένα η φιλοσοφία μα είναι ότι στα πνευμόνια μα τελικά τι καταλήγει και πόσο επιβλαβέ είναι. Αυτό είναι το βασικό. Μία άλλη ερώτηση σε ό,τι το διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τέλη τη δεκαετία του 1990 αναφέρθηκε ότι στι ΗΠΑ υπήρχαν ε, προβλήματα ε, και τότε ήδη είχαν ξεκινήσει επαφέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ για να αποφευχθούν μοναδικά τέτοια σκάνδαλα σε ό,τι αφορά παράκαμψη ε, των ελέγχων. Κοιτάξτε. Ήταν λίγο πριν από τη δική μου την εποχή. Αλλά ξέρω ότι η ομάδα μου δραστηριοποιείται έντονα στις ομάδες εργασίας της Γενέβης. Και τότε η περίπτωση αυτή με τις ε, παραγωγούς ε, μηχανημάτων βαρέων χρήσεων ε, ήταν πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, στην ερώτηση 10 λέει ο κ. Τενές Μάκερ, αναφέρεται τη σύσταση οργάνων για ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συγκεκριμένα λοιπόν σχέδια έχετε σε ό,τι αφορά το δίκτυο αυτό. Χαίρομαι που το έφατε αυτό το ερώτημα. Είναι η απάντηση. Δύο συναντήσεις έχουν συγκληθεί. Τον Απρίλιο ε, έγινε η πρώτη συνάντηση. Τη δεύτερη συνάντηση την διοργάνωσε η Επιτροπή NJRC στην Ίσπρα και η Ιαπωνία, η Κορέα, η Βραζιλία, διάφορα Φυσικά η ΕΠΑ, οι συναδελφοί από την Επιτροπή, όλοι αυτοί συμμετείχαν. Και το συγκεκριμένο σχέδιο που έχουμε είναι το εξή. Να, γίνεται κατά διαστήματα διάλογος, τακτικά διαστήματα, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και εμπειρίες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και την εφαρμογή. Στην τελευταία συνάντηση, λοιπόν, ε, ενημερώσαμε τους συναδέλφους ε, για το που βρισκόμαστε στο θέμα της ε, Volkswagen. Μπεραστήκαμε και διάφορες πληροφορίες για τους ευνηδιαστικούς ελέγχους, κάποια συστήματα για να καταστούν πιο φτηνοί αυτοί οι ελέγχοι, προκειμένου να καταστούν κατά συνέπεια και πιο συχνοί. Θα έλεγα ότι οικοδομούμε σχέσεις και ένα δίκτυο για την ανταλλαγή τακτικών πληροφοριών. Ο κύριος Σάλμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούσα να έρθω στην ώρα μου. Είχε πάρα πολύ ε, κίνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής που θεωρείτε ότι υπάρχουν ε, ισχυρά στοιχεία ε, και ε, που υπάρχουν ασθενή σημεία σε αυτό το πρόγραμμα της Καλιφόρνιας για τα αυτοκίνητα. Λέτε ποια είναι, ποιες είναι οι τάσεις, όχι, όχι, ποιες είναι οι, ποια είναι τα δυνατά σημεία. Εγώ θα έλεγα ότι το δυνατό μας σημείο είναι ότι υπάρχει ένα ε, ε, κεντρικό και πολύ ισχυρό, ε, μια πολύ ισχυρή μάλλον και κεντρική εργαλειοθήκη toolkit που ασχολείται με διάφανο και αποτελεσματικό τρόπο με όλα τα στοιχεία. Και επίσης έχουμε ένα ε, ε, σχέδιο, πρόγραμμα επιβολής και υλοποίησης που είναι διάφανο, αυστηρό ε, και συγκεκριμένο και επίσης ότι ο έλεγχο γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του οχήματο, Όσον αφορά τώρα τα ασθενή σημεία, όπως είπα και προηγουμένως, θα ήθελα ε, να είμαστε λιγότερο προβλέψιμοι από ό,τι στο παρελθόν. Ε, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε, ξεκίνησαμε να το αντιμετωπίσουμε από τον Σεπτέμβριο. Και επίσης εγώ ως ένας, ως ένας μικρός απλός Αμερικάνος λέω ότι κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και επομένως θα πρέπει διαρκώς να αλλάζει και να ε, επικαιροποιείται και να προσαρμόζεται. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να γίνει ένα σύστημα ε, ισχυρό. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπάρχει τέλειο σύστημα. Ερώτηση. Πώς μπορεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία να βελτιωθεί περαιτέρω. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω λεπτομερή γνώση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των προτάσεων που γίνονται στα πλαίσια αυτής. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει ε, μια καλή ε, να υπάρχει καλός συντονισμός, ε, να ε, αλλάζουν οι διαδικασίες έγκρισης τύπου λαμβάνοντας υπόψη ε, τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις και νομίζω ότι ήδη λαμβάνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια άλλη ερώτηση. έχετε ελέγξει οχήματα Chrysler, Fiat, Diesel ε, με την ευρωπαϊκή τεχνολογία απάντηση. Εμείς δεν κάνουμε δοκιμές πάνω σε αυτοκίνητα τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά. Ε, μονάχα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα τα οποία παράγονται για την αμερικανική ε, αγορά αλλά έχουμε ελέγξει ε, BMW, Jaguar ε, και έχουν πετύχει τη διαδικασία έγκρισης τύπου. Εσείς ε, έχετε κάποιες περιπτώσεις όπου η διαδικασία ομολογοποίησης δεν έχει πετύχει. να σας θυμίσω πριν απαντήσω ότι μονάχα πέντε αυτοκινητοβιομηχανίες ε, πουλούν αυτοκίνητα στην, ε, ε, στην Αμερικανική αγορά. Επομένως οι άλλοι γίνονται για BMW, ε, General Motors, Jaguar. Lamborghini. Ερώτηση. έχετε βρει κάποιες ε, ε, περαιτέρω ανομαλίες όσον αφορά τις εκπομπές αυτών των αυτοκινήτων. Ε, απάντηση. Δεν είμαι ακόμα σε θέση να απαντήσω. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμασίες. ο κύριος Άλβα, ελπίζω ότι όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σας θα μπορέσετε να μας απαντήσετε. Ναι, βεβαίως θα το κάνω. Thank you. It's nice to have you Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι εδώ ε, έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη φρασεολογία που χρησιμοποιήσατε. Μιλήσατε για unpredictable tests, για πρόβλεπτες ε, διοδοκιμές. Έτσι όπως τα λέτε, όλα ακούγονται πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει λόγος για πολύ προχωρημένες γνώσεις ε, ε, και τεχνολογικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς ε, πώς γίνονται οι δοκιμές αυτές. Όμως, μια υπηρεσία η οποία είναι τόσο προχωρημένη η δική σας θεωρείτε ότι είναι ένα μάτσο βλακές και δεν μπορέσανε να κάνουν αυτά τα τεστ καλά. Ερώτηση. Ποια ήταν ακριβώς η ερώτησή σας. Δεν την καταλάβατε. Εάν υπάρχει μία οργάνωση, λοιπόν, επαναλαμβάνω, που σύμφωνα με τις γενικές γνώσεις θα μπορούσε να οργανώσει αποτελεσματικά τεστ και δεν το κάνει. Δεν θα το έκανε γιατί είναι ανίκανοι ή γιατί δεν θέλουν να κάνουν αυτά τα τεστ. Ποια είναι η άποψή σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ τώρα να ε, απαντήσω σε μια τόσο υποθετική ερώτηση, γιατί θα ήταν υποθετική και η απάντησή μου, άρα δεν απαντώ. Όμως, στην παρέμβασή σας ε, ε, είπατε ότι οι ευρωπαϊκές δοκιμές ε, είναι γενικώ μη ικανοποιητικές, άρα λέτε εμέσως ότι δεν κάνει τη δουλειά της η Ευρώπη. Απάντηση, όχι. Κοιτάξτε, εγώ μακριά από μένα οποιαδήποτε κατηγορία ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ένα μάτσο βλάκες. Ε, ενδεχομένως δεν χρειάζεται αστροφυσική ε, ε, γνώσης αστροφυσικής ή οτιδήποτε, αλλά παρόλα αυτά ε, χρειάζεται κάτι παραπάνω από το RDE. Οπωσδήποτε χρειάζονται καλά εργαστήρια, χρειάζονται μηχανικοί οι οποίοι να γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους, οι οποίοι επίσης να γνωρίζουν να θέτουν τα σωστά ερωτήματα. Πρέπει να σας πω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, ε, στο ξεκίνημα της διαδικασίας έγκρισης τύπου ε, πρέπει οι κατασκευαστές να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρέπει να αποκαλύψουν κάποια στοιχεία. Αυτό γίνεται πριν. Όταν πουληθεί το αυτοκίνητο τώρα, και το είπα και προηγουμένως, γίνονται άλλου είδους δοκιμές. Γιατί εάν ε, κάποιος κατασκευαστής δεν εξομολογηθεί το αμάρτημά του μόνος του και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε τέτοιες εξομολογήσεις είτε τώρα είτε στο μέλλον, θα πρέπει κανείς σαν η υπηρεσία να είναι ε, σε ε, θέση να κάνει ε, αυτές τις ε, ερωτήσεις ε, ή θα πρέπει να γνωρίζει και θα πρέπει να ξέρουμε τον των προτέρων με ποιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφερθεί το όχημα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, συνθήκες και χρονολογίες. Και αυτές τις έρευνες και αυτές τις δοκιμές ακριβώς κάνουμε και η υπηρεσία της ε, Καλιφόρνια αυτό προσπαθεί να κάνει ε, και μέχρι να πάρουμε ικανοποιητικές απαντήσεις συνεχίζουμε και ε, βελτιστοποιούμε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να φύγω από εδώ και να έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Βεβαίω χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη, χρειάζεται φιλοδοξία, χρειάζεται περιέργεια, αλλά χρειάζεται φυσικά και ο κατάλληλο εξοπλισμό. Και ενδεχομένως και η πολιτική βούληση. Και η βούληση. Ναι, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να θέτει κανείς τα σωστά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Ε, πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε έτσι ώστε να φτάσετε και να αναπτύξετε αυτό ε, το σύστημα δοκιμών. We've working on uh, technology for many, Κοιτάξτε, εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε ε, την ε, επιστήμη των μετρήσεων ε, ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 90. Ξεκινήσαμε κάνοντας ένα σύστημα το οποίο αφορούσε τα βαρέα οχήματα, φορτηγά κλπ. Και σιγά σιγά φτάσαμε ε, στα τωρινά, στις τωρινές δοκιμές. Δεν ε, έχουμε επίσης ε, κάποιο θεσμοθετημένο ως μοναδικό και ενιαίο τεστ. Κάνουμε μία σειρά δοκιμών. Και βεβαίως δεν ρωτάμε και τους κατασκευαστές την άποψή τους, δεν είναι πολύ καλή ιδέα αυτό. Η πρώτη προσέγγιση αφορούσε τα εμπορικά ε, οχήματα ε, και ε, ξεκινήσαμε με αυτές τις μεγάλες υποθέσεις διευθέτησης και συμφωνίας που ακριβώς αφορούσαν περιπτώσεις παραβίασης ε, της νομοθεσίας ε, για τη μόλυνση του αέρα. Ζητήσαμε από τη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει ε, τις συσκευές, αλλά εμείς έχουμε το δικό μας σύστημα επιτήρησης το οποίο λειτουργήσε για τα βαρέα οχήματα και το οποίο τώρα θα διευρυνθεί, όπως είπα και προηγουμένως. Και τι θα λέγατε δηλαδή προς τους Ευρωπαίους αυτοκίνητο ε, βιομηχάνους θεωρούν ότι 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο είναι αδύνατο να το, να το πετύχουμε και πώς πιστεύετε Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο. Ε, πιστεύετε ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να παίζουν κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, η EPA δεν θέτει προδιαγραφές ε, που θεωρεί ε, ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν. Είναι φιλόδοξη και επιθετική ως προς αυτό, αλλά βασιζόμαστε στην τεχνολογία και στα, στα στοιχεία της τεχνολογίας και δίνουμε τη δυνατότητα κάποια χρονική, κάποιο χρονικό περιθώριο στους κατασκευαστές να τα εφαρμόσουν δεν το κάνουμε αυτά στα παρασκήνια. Ε, έχουμε πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα και τα δεδομένα μας είναι όλα στη διάθεση των, ε, ε, του, του, του κοινού. Πιστεύουμε ότι βάσει της νομοθεσίας μας ε, περί καθαρού αέρα έχουμε το καθήκον να πιέσουμε την ε, τεχνολογία προκειμένου να προωθήσει. Πολύ συχνά λοιπόν τα προ... οι δεν βασίζονται σε αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά το τι μπορούμε, τι μπορούμε να, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον, ε, αν έχουμε βέβαια την τεχνολογία να το επιτύχουμε με... η χρηματοδότηση είναι από το... εγκρίνεται από το Κογκρέσο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πιστώσεις ε, που ε, συγκεκριμένα ε, πηγαίνουν προς αυτήν την έρευνα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και που μου ε, που βρίσκεται εδώ, λέει ο κύριο Σέικαουτ. Απλώ ε, θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερο, περισσότερα σε σχέση με την έρευνα και βλέπω και τι γραπτέ ε, απαντήσει από την ΚΑΡΜ, από την Επιτροπή Αερίων Πόρων τη Καλιφόρνια. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώ σα οδήγησε αυτό στην υπόθεση Volkswagen, γιατί από ό,τι κατάλαβα αναφέρονται στο κοινό κέντρο ερευνών και του επενούν γιατί διαφώτισαν ε, και βοήθησαν ε, τους, ε, την Επιτροπή αυτή κάτι το οποίο οδήγησε στην ανακάλυψη της υπόθεσης Volkswagen. Πώς ε, οδηγηθήκατε λοιπόν στο να διερευνήσετε τη Volkswagen. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι συνάδελφοί μου στην Καλιφόρνια ε, και εμείς ε, έχουμε μια πολύ μακρά παράδοση κοινή εργασίας. Είναι κάτι το οποίο ε, έγινε ακόμη πιο έντονο μέσω αυτής της εμπειρίας. έχω στην Επιτροπή αυτή πάρα πολύ καλούς συναδέλφους εδώ και πολλά χρόνια. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό το θέμα της τεχνολογίας diesel, diesel γιατί συνδέεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν ξέρω ακριβώς τη φύση του συντονισμού μεταξύ τους. Ε, μπορώ πάντως να σας πω ε, σε σχέση με την υπόθεση ε, Volkswagen όταν η EPA και η CARB, η Επιτροπή αυτή αερίων πόρων της Καλιφόρνιας έλαβε τα στοιχεία που έδειχναν υψηλές εκπομπές κατά τη χρήση του οχήματος, ε, η Καλιφόρνια αμέσως άρχισε να το ερευνά, έκαναν τις δικές τους ε, δοκιμές, εμείς συμμετείχαμε σε όλες τις, τις ε, συνεδριάσεις ε, λάβαμε, μάλλον κάναμε κάποιες ερωτήσεις, δεν λάβαμε ικανοποιητικές ε, απαντήσεις. Αυτό όμω που άρχισε ουσιαστικά την διαδικασία ε, επιβολής είναι ότι όταν στη Δυτική Βιρτζίνια έγιναν κάποιες δοκιμές αρχικά βασιζόμασταν κυρίως στο θέμα των εκπομπών επομένως υπήρξαν κάποιες διαφορές μεταξύ των εκπομπών που εμείς, που η Volkswagen διατηνόταν ότι υπήρχαν και τις πραγματικές εκπομπές. Ε, έχετε κάποια περισσότερα στοιχεία για τις διατάξεις αναστολής που χρησιμοποιήθηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για το ερώτημα αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η, υψηλού επίπεδου ε, εκπομπές αερίου σε χρήση όταν το όχημα κινείται ε, στο δρόμο και ε, άλλο είναι η διάταξη ε, το, της αναστολής. Μπορεί να είναι ένας ελαττωματικός καταλήτης, ας πούμε, πολύ συχνά κάνουμε ανάκληση οχημάτων για αυτό το λόγο στι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα για να, φανταστούμε και να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για διάταξη αναστολή χρειάζεται πολύ πιο εσβάθο έρευνα ε, πρέπει να είναι κανεί πολύ πιο απρόβλεπτο, ε, να μην ε, ε, βασιστεί τόσο σε εργαστηριακές δοκιμές αλλά σε ε, πραγματικές συνθήκες οδήγησης για να δει κατά πόσο ένα όχημα είναι σχεδιασμένο να συμπεριφέρεται διαφορετικά στον πραγματικό κόσμο από ό,τι σε συνθήκε δοκιμών. Ε, αυτό βέβαια ε, χρειάζεται συγκεκριμένο εξοπλισμό και εμπειρία. Ναι, όμως αυτό υπάρχει και στο Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι λέτε και έχετε και καλές επαφές μαζί τους. Οπότε αν ο κόσμος πει στην Ευρώπη ότι δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία διάταξης αναστολών, εσάς τι σας οδήγησε από τη στιγμή που είχατε από το ICCT τα ίδια ε, στοιχεία από ό,τι και το κοινό κέντρο, ό,τι και όπως, και το κοινό κέντρο Να σας πω ποια είναι η δική μου εμπειρία. Ε, εμείς εγώ και το προσωπικό μου δεν δεχθήκαμε ότι τα, όχημα, τα οχήματα πρέπει να εκπέμπουν ε, περισσότερες εκπομπές ε, χοδρόμο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, από ότι εργαστηριακά. Κάναμε κάποιες ερωτήσεις, δεν λάβαμε ικανοποιητικά από απαντήσεις, ικανοποιητικές απαντήσεις. Αυτό λοιπόν σας οδήγησε, λέει ο κύριος out. Τι σας οδήγησε στο να σκεφτείτε ότι αυτές οι διαφορές ε, δεν ε, ήταν ε, λόγος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αρχίσει η έρευνα δεδομένου ότι τα ίδια δεδομένα, η ίδια εμπειρογνωμοσύνη είναι διαθέσιμη και εδώ. Θα σα πω, λέει ο κύριο Κρούντλερ, κανένα στι ΗΠΑ δεν εξεπλάγει όταν διάβασε την έκθεση ε, του 2009 και 2010 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Εμείς ε, είχαμε αποδώσει αυτές τις υψηλές εκπομπές ε, στις καθόλου, απαιτητικές, καθόλου απαιτητικούς νέους κύκλους δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταχύτητα, επιτάχυνση και δεν γίνεται η δοκιμή επίση στο εργαστήριο υπό διαφορετικέ θερμοκρασίε. Οι περισσότεροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτέ οι διαφορέ ήταν αποτέλεσμα του κύκλου δοκιμών και όχι ε, επειδή κάποιο πήρε εσκεμένα την απόφαση να, ε, κλέψει. Αυτή ήταν ε, η απόφαση μα τότε και βεβαίω έγιναν και πάρα πολύ σοβαρέ δοκιμέ υπό τον δικό μα κύκλο δοκιμών. Κάτι το οποίο είναι επίση πολύ σημαντικό είναι ότι το ε, ε, όχημα το οποίο δημιουργείται για την αμερικανική αγορά είναι πολύ διαφορετικά από τα 5-6 που κατασκευάζονται εδώ, γιατί είναι διαφορετικά σε προδιαγραφές ε, είναι πιο απαιτητικέ οι προδιαγραφέ, πιο απαιτητικοί οι κύκλοι δοκιμών, ε, τα οχήματα diesel που πολλούνται στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλότερε προδιαγραφέ και να μπορούν να περάσουν έναν πολύ πιο απαιτητικό έλεγχο. Γι' αυτό ακριβώ εμεί δεν σκεφτήκαμε ότι, μας, ότι ήταν περίεργο αυτό, γιατί οι προδιαγραφέ είναι διαφορετικέ, τα οχήματα είναι διαφορετικά και ε, οι κύκλοι δοκιμών είναι διαφορετικά. Η κυρία Εύη. Θα σας τα πω στα Ιταλικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την απάντησή σας στην ερώτηση περίπου 10 όπου λέγεται ότι η EPA συμμετείχε στο νέο κύκλο ε, δοκιμών για τις διαδικασίες ε, έγκρισης ε, τύπου έτσι ώστε να βελτιωθούν οι ελλείψεις του, της, της ευρωπαϊκής πρότασης. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι, κάποιες, κάποια, ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι ώστε να λαμβάνετε υπόψη υπόψη η χρήση ε, των οχημάτων και κατά την άποψή σας γιατί οι ευρωπαϊκές αρχές ε, δεν ε, έλαβαν τέτοια μέτρα όσον αφορά το, τις παγκόσμιες εναρμονισμένες αρχές, γιατί δεν συμμετέχετε πλέον, γιατί δεν ακολουθείτε αυτό το τεστ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Ναι, συμμετείχαν και μέλη της δικής μας ομάδας στις συναντήσεις ε, στη Γενέβη. Δικός μας ρόλος λοιπόν ήταν να παράσχουμε τα δικά μας, ε, τις δικές μας εμπειρίες σε ό,τι αφορά τους κύκλους αυτούς δοκιμών και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που ισχύει σε μας. Αυτό μάλιστα έγινε μετά τις εκλογές ε, τις τελευταίες της είπα. Και η ομάδα μου είχε λάβει την εντολή από τον πρόεδρο Ομπάμα τότε να ξεκινήσει τις εργασίες για την ανάπτυξη τέτοιων προτύπων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Άρα χρειάστηκε να δώσουμε προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την πολιτική και έτσι να δημιουργηθεί το πρώτο πρότυπο για το διοξείδιο του άνθρακα για τις ΕΙΠΑ. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο δέσμευση και συμμετοχής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Θεωρούμε ότι οι πέντε κύκλοι είναι υπερισχύουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύστημα. Προφανώς δεν πείσαμε γιατί το WLTP δεν περιλαμβάνει όλα όσα περιλαμβάνονται στους πέντε κύκλους και εμείς δεν προτιθέμεθα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε την νομοθεσία μας ε, για μια νομοθεσία η οποία δεν ε, είναι εξίσου καλή. Αυτό καταρχάς και κατά δεύτερον η προσαρμογή του κύκλου δοκιμών στη μέση της διαδικασία ε, παραγωγής θεωρώ ότι θα ήταν επιβλαβής και για την βιομηχανία και για τον απότερο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε που είναι η μείωση των εκπομπών. Ε, Σας ευχαριστώ. Μια άλλη ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, η EPA ε, διεξάγει τα τεχνικ, τις τεχνικές δοκιμές πριν ε, τα οχήματα μπουν στη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή ελέγχει και τα πρωτότυπα. και εσείς κάνετε, εσείς ζητάτε και τις δικές τους δοκιμές, αυτές που κάνουν in-house ε, ή και από, ε, από τις ε, ειδικές, από τις, συγγνώμη, από τις ιδιωτικές ας πούμε εταιρείες ή όλα τα κάνετε εσείς. Η απάντηση είναι ναι. Πώς γίνεται οι κατασκευαστές πρέπει να κάνουν τις προδιαγραμμένες δοκιμές στα εργαστηριά τους. Κάποιοι μπορούν να το αναθέσουν, αλλά οι μεγάλες εταιρείε έχουν δικιά του τμήματα. Μας στέλνουν στη συνέχεια τις πληροφορίες αυτές, τα στοιχεία αυτά, στα πλαίσια των αιτήσεων για την έγκριση και στη συνέχεια κάνουμε έναν έλεγχο σε 20-30% των καινούργιων αυτών οχημάτων γίνεται μια εντολή ε, δοκιμών και μας παραδίδουν το όχημα στα εργαστηριά μας και εκεί κάνουμε τους δικούς μας ελέγχους, τις δικές μας δοκιμές. Αν καταλήξουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα από ότι οι κατασκευαστές υπερισχύει το δικό μας πόρισμα, το δικό μας αποτέλεσμα και βάσει αυτού αποφασίζεται κατά πόσον πληρούνται ή όχι οι προδιαγραφές για το όχημα. Επίσης ελέγχουμε τα, τα οχήματα που προέρχονται από τη γραμμή παραγωγής. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στον κατασκευαστή ή να τους πούμε να μας στείλουν ένα όχημα από τη γραμμή παραγωγής και να κάνουμε σε αυτό το έλεγχο, να δούμε κατά πόσον δηλαδή είναι το ίδιο με το πρωτότυπο, το πρότυπο που έχουμε ελέγξει και επίσης ε, χρησιμοποιούμε και διάφορες ε, πηγές από τους πολίτες. Ο κύριος Μπελέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γκρούντλερ ε, που είναι μαζί μας και συγγνώμη που θα σας θέσω την εξή ερώτηση. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις για το σκάνδαλο για τα αυτοκίνητα diesel στο, στη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά τα τεράστια πρότυπα, την πολύ αυστηρή αντιμετώπιση των κατασκευαστών και αυτό εξετάστηκε από πλευράς ανταγωνιστικότητα. Τα τεράστια λοιπόν αυτά πρότυπα αναφέρθηκε ότι είχαν ε, μάλλον οικονομικό υπόβαθρο για να καταστήσουν την πρόσβαση στην αμερικανική αγωγή, αγορά πιο δύσκολη στους ξένους παραγωγούς και ιδιαίτερα στους παραγωγούς ε, αυτοκινήτων diesel. Πώς το σχολιάζετε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, λέει στην απάντηση ο κύριος Ε, δεν συμφωνώ προφανώς με την ε, ανάλυση αυτή. Υπάρχουν σαφή μητρώα τα οποία δημοσιεύονται Να κοιτάξουν λοιπόν οι αναλυτές τα σχετικά μετρώα για να κρίνουν κατά πόσον συμβαίνει αυτό ή όχι. Σε ό,τι αφορά την αυστηρή αντιμετώπιση, να πω ότι ποτέ δεν έχουμε δει μια τέτοια περίπτωση στην ιστορία μας ότι ο υφυπουργός μας, ο, μάλλον ε, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ίδιο δήλωσε σε ό,τι αφορά πρόστιμα, να σας πω ότι δεν έχουμε αξιολογήσει το ύψος των προστήμων έως τώρα. Μια μερική διευθέτηση έχει ανακοινωθεί, η οποία και αυτή ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και στην παρούσα φάση δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Πέρα από το ότι το θέμα των ε, μερικών διευθετήσεων έχει να κάνει με το χημά, έχει να κάνει και με την βλάβη που προκληθήκε στο περιβάλλον. Δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί τα θέματα προσθήμων. Ναι, σύμφωνο, αλλά κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία, το σκάνδαλο πριν από 20 χρόνια είχε να κάνει με τα βαρέα οχήματα. Ένα δισεκατομμύριο έως και 15 δισεκατομμύρια αναφέρεται το ποσό των προστήμων. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες αποκλήσεις. Αυτό ενδεχομένως να οδήγησε στην συγκεκριμένη ανάλυση. Κοιτάξτε, οι αναλύσεις αυτές πολύ απλά είναι ασφαλμένες. Δεν ε, είχαν εκτιμηθεί τα πρόστιμα, άρα πώς να γίνει σύγκριση τιμών. Τα ποσά που αναφέρεται έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, των οχημάτων. Γιατί τα οχήματα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν συμβατά στη ΣΥΠΑ. Και άρα ο αγοραστής ή θα επιστρέψει το όχημα ή θα πάρει μια τροποποίηση των εκπομπών του. Και τα οχήματα λοιπόν αυτά, αν παραμείνουν στον δρόμο, Ε, μάλλον τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν και την βλάβη που προήλθε από την εκπομπή των αζωτούχων, των νόξ και φυσικά έχουν να κάνουν και με τις επενδύσεις που έχει συμφωνήσει να κάνει η Volkswagen σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μελλοντικής τεχνολογίας. Εδώ δεν έχουν εκτιμηθεί δηλαδή πρόστιμα. Ναι, γιατί πολύ απλά όταν βγάζει στην αγορά 600.000 προβληματικά αυτοκίνητα, αυτό έχει κόστος. Είναι λογικό. Ευχαριστώ, κύριε Ντάλη. Έχει το λόγο. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρούντλερ που βρίσκεται εδώ μαζί μα και που μα ε, δίνει τις πληροφορίε αυτές. Δύο σημαντικά στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω από την παρουσίασή σας στο θέμα των επενδυαστικών ελέγχων και το γεγονός ότι διαρκώς πρέπει να τροποποιείται τις δοκιμές που κάνει η EPA. Γιατί το θέμα λοιπόν αυτό και όλος ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά και την γραπτή απάντηση στην ερώτηση 5, αναφέρεται ότι η EPA δημιούργησε νέες διαδικασίες ελέγχων για τα βαρέα και τα ελαφριά οχήματα, προκειμένου να α, τηρούνται τα πρότυπα. Όταν γίνεται όμως αναβάθμιση τέτοιων δοκιμών, ε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αυτό πρέπει να γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς να υπάρχει να χρονοτρεβεί κανείς. Πόσο καιρό λοιπόν πήρε η εφαρμογή του νέου καθεστώτος δοκιμών από πλευρά της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο καιρό παίρνει αυτή η αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλές ερωτήσεις σας. Ε, προσαρμόσαμε τις ε, πρόσθετες ομοσπονδιακές διαδικασίες όπως σας αναφέρουμε το 1996. Και έτσι εφαρμόστηκαν το 2000. Μας πήρε χρόνο λοιπόν. Μας πήρε χρόνο να προσαρμοστούν αυτές οι διαδικασίες ε, πρόσθετων δοκιμών. Το 2000 λοιπόν εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ και εφαρμόστηκαν και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διευθυντήτου του άνθρακα σε τη φατάρια θερμοκηπίου. Κοιτάξτε, δεν είναι και μικρή δουλειά να εγκριθεί μια νέα διαδικασία ελέγχου και ακολουθήσαμε και μια δημόσια διαδικασία με συμμετοχή και της βιομηχανίας και των εμπειρογνωμόνων. Πήρε χρόνια λοιπόν, ναι, αλλά πόσο πήρε όλη η διαδικασία, λέει η κυρία Νταλή. Είπατε ότι συμμετείχε και η κοινή γνώμη. Κοιτάξτε, απάντηση. Τι ήθιστε. Τελευταία. Μας παίρνει ένα-δύο χρόνια η ανάπτυξη μιας νέας πρότασης. Ανάλογα και από το πεδίο εφαρμογή της ρυθμιστικής πρότασης. Και 12 μήνες μας ε, παίρνει, ένα χρόνο δηλαδή, η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και αριστικοποίησης της διαδικασίας και των προτύπων, η Νταλή. Ναι, αλλά παράλληλα καταφέρνετε να διατηρείτε και τον παράγοντα των ευνηδιαστικών των ελέγχων, των απρόβλεπτων ελέγχων, για να διασφαλίσετε ότι η εργαστηριακή εκπομπή είναι η ίδια με την πραγματική. Κοιτάξτε, είναι νέο στοιχείο αυτό η απάντηση. Αλλά όπως σας είπα, στο τέλος της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν αυτές οι διαδικασίες και είχαν πάρει και χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον απρόβλητο χαρακτήρα των ε, διαδικασιών, αυτά εφαρμόζονται σε 24 ώρες. Μόλις δηλαδή καταρτίστηκε το σημείωμα παραβίασης και επειδή έχουμε μάθει και το μάθημά μας σε ό,τι αφορά το απρόβλεπτο του συστήματος, στέλνουμε μια επιστολή λοιπόν στον παραγωγό, όπου του λέμε με την αρμοδιότητα και τις ε, εξουσίες που έχουμε, σας ζητούμε να κάνετε εσείς τον έλεγχο ή θα το κάνουμε εμείς τον έλεγχο. Μάλιστα. Αυτό το κριτήριο λοιπόν, το ευνηδιαστικό, μπορεί να αλλάξει, να προσαρμοστεί σε 24 ώρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλη χρονική διάρκεια. Ναι, γιατί έχουμε πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα εργαλεία στα πλαίσια της νομοθεσίας για την καθαρή ατμόσφαιρα. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι τα οχήματα πρέπει να πληρούν τους ε, πρότυπα εκπομπών σε όλες τις φυσιολογικές καταστάσεις λειτουργίας. Και επίσης ε, η νομοθεσία μας δίνει την αρμοδιότητα να ελέγχουμε ανα πάσα στιγμή όπου θέλουμε όποιον κατασκευαστή θέλουμε, υπό κάποιους όρους βέβαια. Για παράδειγμα, ζητήσαμε από ένα συγκεκριμένο παραγωγό να ελεγχθεί ένα όχημα σε διάφορες δημοκρασίες και να μας υποβάλει τις πληροφορίες αυτές ε, στην υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε μαθητική διαδικασία για να επιβληθεί μια νέα μορφή δοκιμών η Και αυτό ίσως να είναι το κλειδί που σας επιτρέπει, αυτό μπορεί να σας επιτρέπει να μην έχετε παραγωγούς που να υποσκάπτουν το σύστημα. Ναι, θα έλεγα ότι αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς, γιατί από πέρσι το Σεπτέμβριο δεν ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο γίνεται ο έλεγχος. Κοιτάξτε, κάποιες ερωτήσεις για το σύστημά σας. Όταν ε, η EPA ε, κάνει τέτοιες ελέγχου σε ιδιωτικά οχήματα, είναι προφαντικό αυτό ή φρεντικό. Και επίσης πείτε μας, η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος ε, ε επιβάλλει τέλη στους παραγωγούς για την διεξαγωγή των δοκιμών και την πιστοποίηση. Πώς, ε, σε ποια βάση λοιπόν επιβάλλονται τα τέλη αυτή, βάση των πολλών οχημάτων ή πώς τι ιδιώτε προσλαμβάνουμε. Κοιτάξτε, είναι θελοντικό. Παίρνουν μια φιλική επιστολή από την EPA που λέει πώ θα θέλατε να συμμετέχετε, να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα ε, δοκιμής ε, για τον καθαρό αέρα. Θα σα δώσουμε ένα νέο και αυτοκίνητο ε, το οποίο θα σα το καθαρίσουμε και θα το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Προσπαθούμε τέλο πάντων να αξίζει το κόπο. Έχουμε συγκεκριμένο, συγκεκριμένη νομοθεσία για, τη, για τα τέλη. Έχει σχέση με τον υπολογισμό του έμεσου κόστους ε, για το πρόγραμμα συμμόρφωσης και για το πρόγραμμα ε, δοκιμών. Ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό, μπορεί να είναι 25.000 δολάρια, για μια συγκεκριμένη οικογένεια ε, οχημάτων, ε, τα συλλέγουμε και τα στέλνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, το Κογκρέσο κάθε χρόνο τη Σοφία το αποφασίζει ποιο θα, ποιος θα είναι ο προπολογισμό της υπηρεσίας μας. Θέλουμε να πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχέση, αλλά δεν είναι πολύ άμεση σχέση. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γκυζίτσκι. Κύριε Γκρούντλερ, ε, έχετε έξι λεπτά και εγώ έχω τρία λεπτά να δούμε την πρώτη ερώτηση που δεν απαντηθήκε σωστά γιατί α, ρώτησα πώς αντιδράει η βιομηχανία στις διαδικασίες αυτές γιατί μας περιγράψατε τι γίνεται με την κοινή γνώμη. Αλλά, για παράδειγμα, η Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε τι βαθμό συμμετέχει επίσημα στη διαδικασία και κατά πόσον συμμετέχουν ε, με ενδιαφέρει και ευρωπαϊκές ε, ε, υπηρεσίες για την προάσπιση των ευρωπαϊκών ε, συμφερόντων. Στο τι βαθμό λοιπόν συμμετέχουν όλοι αυτοί. Συγγνώμη που δεν απάντησα πλήρως. Ε, μιλάω γενικά για το κοινό. Συμμετέχουν οι ε, αυτοκίνητο βιομηχανίες, γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι ετοιμάζουν, τι υπάρχει στο εργαστηριό τους, πώς βλέπουν την ε, αγορά, την τεχνολογία, τι, τι θεωρούν ότι υπάρχει ως δυναμικό για την τεχνολογία. Οπότε συμμετέχουν ενεργά ως προς τη ρυθμιστική μας προσέγγιση. Εμείς πηγαίνουμε συχνά στη Γερμανία, ε, στην Ασία, στο Ντιτρόιτ, ε, σε ε, εγκαταστάσεις όπου η τεχνολογία εξελίσσεται και προσπαθούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες. Κάνουμε λοιπόν και εμείς τη δική μας δουλειά και έχουμε και τα δικά μας εργαστήρια όπου αξιολογούμε τις καινούργιες τεχνολογίες για να μπορέσουμε, για να, για να, μπορέσουμε να ορίσουμε τους στόχους μας για τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου το 2025. Ε, εμείς ε, μπαίνουμε στον εγκέφαλο για να ξέρουμε πώς οι κατασκευαστές ελέγχουν τον εγκέφαλο της μηχανής, για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο στις συνεδριάσεις μας με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες πληροφορίες σε συναντήσεις ένας προς έναν. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι τμήμα της δουλειάς. Ε, και πηγαίνουμε ε, στην δική τους εγκατάσταση, ε, κάνουμε ερωτήσεις στους μηχανικούς τους για να πάρουμε τις πληροφορίες μας. Σας ευχαριστώ. Ικανοποιητική πολύ η απάντησή σας. Μας είπατε επίσης ότι είναι πολύ καλή χρηματοδότηση της υπηρεσίας σας, ότι έχετε υπαλλήλου. Εμείς είμαστε μια ερευνητική επιτροπή που έχουμε απλά συστάσεις να δημοσιεύσουμε για το μέλλον. Επίσης συνεργαζόμαστε με το JRC, το Κέντρο Ερευνών και την ΙΣΠΡΑ. Για τους υπαλλήλου μπορείτε να μας πείτε τι χρηματοδότηση έχετε. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ποιοι ερευνητέ ερευνούν και ποιοι οι ερευνητέ είναι συγκεκριμένα, συμμετέχουν στην, στον έλεγχο, στη δοκιμή. Και κάτι άλλο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερο, επειδή δεν ήταν θέμα hardware, αλλά software η απάτη. Τι εμπειρογνώμονε έχετε για θέματα software, λογισμικού και θα λέγατε ότι είσαστε αυτόνομοι σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη δηλαδή ε, το, της απάτης της Volkswagen σε ό,τι αφορά το λογισμικό το ανακαλύψετε μόνοι σας με τους εσωτερικούς σας υπαλλήλου ή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε και εξωτερικούς. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την εξίσου περιεκτική ερώτηση. Καταρχά εγώ δεν είπα ποτέ ότι το Κογκρέσο μας δίνει επαρκής πόρους. Ε, μας δίνει πόρους ε, και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες ε, για αυτά που επιλέγουν να μας παρέχουν. Στην οργάνωσή μας έχουμε περίπου 350 υπαλλήλους για τις ευθύνες που ανέφερα ε, και για τα καύσιμα και για τα οχήματα, όχι μόνο για τα οχήματα. Από τα 350 άτομα θα έλεγα ότι περίπου 200 και αυτές είναι, τεχνικοί αυτή είναι τεχνική πόρη, δηλαδή ε, δοκιμαστές, ε, μηχανικοί κλπ. οι 200 περίπου έχουν άμεση σχέση με την επίβλεψη της συμμόρφωσης των οχημάτων, των δοκιμών των, των οχημάτων, και περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια που μας βοηθά ε, στη δουλειά μας, ε, στην απόκτηση οχημάτων κλπ. Όλα αυτά γίνονται βέβαια, οι τα περισσότερα ε, από τα τεστ γίνονται εντός της υπηρεσίας μας. Δεν είναι κάτι με το οποίο θα μπορούσαμε να επιφορτήσουμε ένα ιδιωτικό εργαστήριο ή κάποιον ανάδοχο. Όσον αφορά τώρα για το λογισμικό και τους σχετικούς ε, και τους υπεύθυνους. Ε, έχουμε μια διαδικασία ε, πρόσληψης που μας επέτρεψε να ε, προσλάβουμε πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους από την, ε, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που πριν έρθουν ε, στην υπηρεσία μας έκαναν διαμόρφωση λογισμικού προκειμένου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους με, τις συγκεκριμένα, με τα συγκεκριμένα προσόντα που έχουν να κάνουν πούμε, με ένα ελαφριό χύμο. Εγώ, για παράδειγμα, παράδειγμα στην προηγούμενη μου δουλειά έπρεπε να φέρνω ένα ε, ελαφρύ όχημα από ε, το χώρο που σχεδιαζόταν ε, μέχρι την αντιπροσωπή αυτοκινήτου που το πουλούσαν. Χρειάζεται πραγματικά πολύ ταλέντο για να κάνει κανείς αυτή τη ε, δουλειά δεν χρειάζεται να, να, ε, ε, εξετάσουμε εκατοντάδες λογισμικά για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει μια διάταξη αναστολής. Δεν χρειάζεται να περάσουμε από εκατοντάδες κωδικούς μπορούμε να ε, ζητήσουμε στον ε, κατασκευαστή να μας δώσει το κλειδί που ξεκλειδώνει ε, το όχημά του και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς σχεδιάστηκε και πώς κατασκευάστηκε το όχημά του. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ, μια πολύ καλή και ευρία εργαλειοθήκη στη διάθεσή μας, αλλά έχουμε και πόρους αλλά δεν είναι αρκετοί. Άμα ξέρετε κανέναν λοιπόν στο Κογκρέσο και μπορείτε να μας βοηθήσετε, μάλιστα ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία ε, Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και που απαντάτε με τόση ακρίβεια στις ερωτήσεις μας. Ε, εγώ έχω μία ερώτηση σε σχέση με τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ε, που είναι τμήμα των κύκλων δοκιμών που, γίνεται, που κάνετε κι εσείς. Από πότε τις κάνετε αυτές τις δοκιμές και πόσο καιρό χρειαστήκατε για να μπορέσετε να τελειοποιήσετε μία αξιόπιστη τεχνική. We adopted um, εμείς εγκρίναμε την νέα, ε, τους νέους βελτιωμένους κύκλους δοκιμών μας ε, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και ήταν ε, ήδη επιχειρησιακή την, ε, ε εντός της επόμενης δεκαετίας και μιλάω τώρα για τον κύκλο που αφορά τις υψηλές ταχύτητες και αυτά που σας εξήγησα και σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν την ευρεία εμβέλεια των ε, συνθήκων που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα οχήματα. Αυτοί οι πέντε κύκλοι ε, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος κάτω από τους ε, μείον 7 βαθμούς Κελσίου, πάνω από 27 βαθμούς, ε, από 0 μέχρι 100, μέχρι 199, άμεση επιτάχυνση, άμεση επιβράδυνση. Όλα αυτά θεωρούμε ότι ένα απλό και σύνηθες όχημα πρέπει να αντιμετωπίσει ως συνθήκη χρήσης. Δεν μπορώ να σας πω τώρα πόσο χρόνο χρειαστήκαμε. Ε, αυτούς τους τρεις επιπλέον κύκλους, ε, τους, τους τελευταίους που εγκρίναμε, χρειάστηκαν κάποια χρόνια εργασίας. Ο πιο πρόσφατο, στο πιο πρόσφατο ε, δίδαγμα που είχαμε είναι ότι πρέπει να είμαστε απρόβλεπτοι ευνηδιαστικοί κάθε όχημα που ελέγχουμε, όταν βλέπουμε ότι μια διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και επαναλαμβανόμενη, έχουμε μια εργαστηριακή μέθοδο που καλύπτει πάρα πολλές συνθήκες. Είναι σημαντικό να περάσει από, όλες αυτές, ε, από όλους αυτούς τους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια συσκευή, μια διάταξη ε, ε, αναστολής. Επίσης έχουμε και κάποιες κινητές μονάδες στο δρόμο. Δεν θεωρούμε ότι μόνο στο εργαστήριο μπορεί να γίνονται αυτές ε, οι αυτή η έλεγχη χρειάζεται μια πιο περιεκτική προσέγγιση, πιο πλήρης άμα θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα για καθαρότερο αέρα. Οπότε το κάνετε αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δηλαδή περίπου 16 χρόνια περίπου κάνετε τέτοιου είδους σε πραγματικές συνθήκες ελέγχους η νομοθεσία αμερικανική έχει προβλέψει όλα αυτά τα είδη ελέγχου. Ε, σας δίνει λοιπόν ένα μια υποχρέωση αποτελέσματος. Ε, πρέπει να έχετε κανόνες ε, τους οποίους δεν πρέπει να τους ξεπεράσετε ή έχετε στη διάθεσή σας τη διακριτική ευχέρεια που σας επιτρέπει να καταλάβετε ε, τι πρέπει να κάνετε. Η νομοθεσία είναι πολύ ακριβής για τα διάφορα είδη ελέγχων ή εσείς ως Ομοσπονδιακή υπάλληλοι έχετε τη δυνατότητα να την υλοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο που εσείς νομίζετε και όταν θεωρείτε ότι πρέπει να την εξελίσσετε γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται και αυτή, μπορείτε να το κάνετε ή πρέπει κάθε φορά να περνάτε από μία νομοθεσία μπροστά από το ε, Κοινοβούλιο για να το επιτύχετε. Αυτή είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Νομίζω ότι η απαρχή ε, αυτών των νέων πιο απαιτητικών ε, δοκιμών ε, υπήρχε στην νομοθεσία, είναι τμήμα τροποποιήσεων και επιπρόσθετων, επιπρόσθετης νομοθεσίας, της νομοθεσίας του 90 για τον καθαρό αέρα είναι αλήθεια ότι έχουμε κάποιους ε, υποχρεωτικούς ε, ελέγχους ε, που εγκρίνονται από την ομοθεσία, που μας δίνουν τη δυνατότητα, μας δίνουν την ευχέρεια να ελέγξουμε και ε, μέσω ε, κανονικών αλλά και μέσω μη κανονικών κύκλων ελέγχων μπορούμε να προσαρμόσουμε τους κύκλους δοκιμών όπως το κάναμε από το περασμένο Σεπτέμβρη για να ελέγξουμε σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε λογικές συνθήκες τις οποίες ε, θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κανονική του λειτουργία ένα όχημα. Δεν θα ήταν λογικό για μας να κάνουμε ε, μία δοκιμή σε 120 βαθμούς Φαρενάιτ ε, γιατί πολύ σπάνια θα βρεθεί ένα όχημα σε τέτοιες ε, θερμοκρασίες όμως 85 βαθμοί Φαρενάιτ ναι 35 βαθμοί Κελσίου δηλαδή ε, είναι λοιπόν ε, πραγματική μας ε, προσδοκία ότι θα έπρεπε κάποιες προδιαγραφές να γίνονται σεβαστές υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και έχουμε κάποιες εκ του νόμου υποχρεώσεις δοκιμών, κύκλων δοκιμών και έχουμε και, κάποιες άλλες, και κάποιες άλλες μεθόδους τις οποίες τώρα δεν θα σας περιγράψω. Μία ακόμη ερώτηση, πολύ σύντομα θα είδατε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ε, αυτοκινητοβιομηχανίες ε, ε, που σταματούν την έκκληση οξυδίων του αζότου πέρα από κάποιες θερμοκρασίες από μείον 7 έως τις 35 εσείς θεωρείτε ότι είναι μια κανονική λειτουργία. Εσείς ποια είναι, η αποψή σας για αυτήν την προσέγγιση και αυτήν τη στάση των Ευρωπαίων ε, αυτοκινητοβιομηχάνων. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας ε, μετριόφρον ε, Αμερικανός. Ε, πράγματι, έχουμε πολύ, μια πολύ μεγάλη γκάμα και αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της ρυθμιστικής μας ε, προσέγγιση στο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας μας. Είναι λογικό να θεωρήσει κανείς ότι στην Αμερική θα, έπρεπε, θα αντιμετώπιζε κάποιε τέτοιε συνθήκε από μείον 7 βαθμού Κελσίου μέχρι 35 ένα όχημα στην Αμερική. Ε, γι' αυτό έχουμε ακριβώ τόσο ευρεία κλίμακα ε, θερμοκρασία. Γι' αυτό ακριβώ εγκρίναμε το RDE, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Κύριε Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκρούντλερ, είπατε προηγουμένω ότι σε ό,τι ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το RDE αποτελεί ένα βήμα προς τη κατεύθυνση. Το θέμα όμως είναι ένα πραγματικά επαρκής και να αναφέρω και τους παραγόντες σημαντότητας. Στις ΗΠΑ γνωρίζουμε ότι ο παράγοντας, ο συντελεστής ε, συμβατότητας είναι 0,4. Πώς το αξιολογείτε λοιπόν αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω ε, σε τι αναφέρεστε σε ό,τι αφορά το συντελεστή συμβατότητας συμμόρφωσης 0,4. Δεν το γνωρίζω. Εκτός αν αναφέρεστε στο όριο που δεν πρέπει να ξεπερνέτε από τις ε, βαρέους κινητήρες. Ε, δεν υπάρχει τέτοιο συντελεστής όμως για τα επιβατικά. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή συντελεστή συμμόρφωσης, αν κατάλαβα σωστά, λέει ο κ. Δεμέσμακερ. Ε, μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω. Μήπως δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Να απαντήσω το εξής. Ε, τα οχήματα εν λειτουργία περιμένουμε να έχουν τα ίδια αποτελέσματα από τα εργαστηριακά. Χρησιμοποιούμε συσκευές εντοπισμού των προβλημάτων. Αν βρεθούν λοιπόν τα, αν εντοπιστούν προβλήματα, χρησιμοποιούμε και την εργαστηριακή και τις άλλες μεθόδους, αλλά οι εκπομπές πρέπει να είναι παρόμοιες. Δεν θα είναι ποτέ ταυτόσιμες. Προφανώς γιατί αλλάζει διαρκώ ο πραγματικός κόσμος, αλλά θα πρέπει να είναι παρόμοιες. Αν δεν είναι παρόμοια τα αποτελέσματα, υπάρχει πρόβλημα. Οχήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο δρόμο από ότι στην, στο εργαστήριο, τα θεωρούμε διατάξεις αναστολής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την ίδια προσέγγιση σε ό,τι αφορά το RDA. Χρησιμοποιείται αυτό σαν μηχανισμός έγκριση τύπου. Εμεί ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση και θα παρακολουθούμε διαρκώς τις εμπειρίες σας με το RDE και προφανώς θα προσαρμόσουμε τη διαδικασία μας εάν θεωρήσουμε ότι αυτό ενδείκνεται αλλά δεν έχω άποψη εδώ και τώρα, σήμερα, να σας παρουσιάσω σε ό,τι αφορά το συντελεστή συμμόρφωση, αν είναι επαρκή ή όχι, γιατί πολύ απλά δεν έχω επαρκή στοιχεία στη θέση μου. Λυπάμαι. Μάλιστα. Η κυρία Κιλιόναν. Σας ευχαριστώ για το δεύτερο γύρο να μιλήσω αγγλικά. Εκπροσωπώ την ΚΟΥ λοιπόν και νομίζω ότι εδώ ε, στην Ευρώπη ε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προστατεύουμε τη βιομηχανία, της εταιρεία. Ξεχνάμε όμως τον ε, πελάτη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς, με την εκτίμησή σας, πιστεύετε ότι η νομοθεσία σας για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι πιο σωστή και αντεκνιόμενη σε σχέση με την ευρωπαϊκή και πώς βλέπετε το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας γιατί η κατάσταση στην αγορά είναι αρκετά ζωφερή στη ΣΥΠΑ από ό,τι κατάλαβα. Πώς ε, θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του Αμερικανού καταναλωτή σε ό,τι αφορά και την τεχνολογία diesel. Πώ εκτιμάτε λοιπόν την κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση την οποία και τέτοιτε. Δεν είμαι ειδικό στην προστασία του καταναλωτή και τέτοια θέματα που άπτονται προστασία τη προστασία του καταναλωτή τη ΕΠΑ. Εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε ε, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις για τις εκπομπές. Και η Volkswagen είχε συμφωνήσει να κάνει κάποιες τέτοιες τροποποιήσεις. Η διευθέτηση ήταν σε συνάρτηση και με τις αρχές προστασίας του καταναλωτή της είπα. ΕΕ. Αυτές ήταν οι υπεύθυνε. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικό για θέματα που άπτονται του σκέλους της προστασίας του καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά το μέλλον τώρα του κλάδου, να κάνω κάποια σχόλια. Είπατε ότι ήταν δύσκολο. Δεν είμαι και βέβαιος. Η αυτοκινητοβιομηχανία στη ΣΥΠΑ δεν τα πάει καθόλου άσχημα. Ανθεί. Τρία χρόνια πολύ καλές πωλήσει. Το 2015 ήταν έτος ε, ρεκόρ. Έξι συναπτά έτη αύξηση των πωλήσεων, να σας πω. Και οι μαρικανικοί κινητέρε έχουν ε, τις πιο πολλές δυνατότητες της αγοράς και ιδιαίτερα τα φορτηγά και τα SUV ε, έχουν ωφεληθεί όλος ιδιαίτερος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα για τα για τις ε, εκπομπές θερμοκηπίου τα πηγαίνει φανταστικά. Μην σας πω ότι η παραγωγή υπερβαίνουν τα πρότυπα αυτά. Και πιστεύω ότι και μετά το 2025 θα παραμείνουν ενδιαφέρουσες ε, οι ισορροπίες αυτές. Τώρα για τα δίζελ είναι ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό. Γιατί προφανώς έχει πληχθεί το κύρος των δίζελ στην Αμερική. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν βασικά φορολογικές, ε, φορολογικοί λόγοι. Καταρχάς δεν υπάρχει διαφορά στην φορολογία στην Αμερική, δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος να επιλέξει κανείς δίζελ. Υπάρχει φυσικά πλεονέκτημα στην αποδοτικότητα, όχι όμως φορολογικά. Και το δίζελ αντιμετωπίσει φυσικά ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την προηγουμένη ε, βενζίνη και τα ευρυδικά. Νομίζω λοιπόν ότι ο όμιλος Volkswagen πολλούσε τη μεγάλη πλειονότητα, το μεγαλύτερο κομμάτι των δίζελ στην Αμερική. οι Mercedes ε, και η BMW μόνο μικρό μερίδιο της αγοράς diesel είχαν. Άρα πιστεύω ότι είναι θέμα της αγοράς πιο πολύ. Οι Αμερικανοί οδηγοί θυμούνται ε, ακόμα καλά τις πρώτες κινητήρες diesel της General Motors που ήταν ε, πάρα πολύ, έτσι, πώς να πω, ε, δύσκολη εμπειρία. Ήταν βρώμικοι κινητήρες, Και πρόσφατα πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε κατά τον δίζελ, είμαστε υπέρ του καθαρού αέρα, της καθαρής ατμόσφαιρας. Ε, προσφάτως, μάλιστα, εγκρίναμε και τρία νέα οχήματα. Άρα πιστεύω ότι θα φανεί με την πάροδο του χρόνου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και κατά πόσον θα ξανακερδίσει το δίζελ τον καταναλωτή. Ξέρουμε ότι πολλοί καταναλωτές που θέλουν να πουλήσουν δίζελ στη ΣΥΠΑ Jaguar Land Rover για παράδειγμα. Και τα δύο αυτά, και δύο αυτοί όμιλοι έχουν εντελώς νέα προϊόντα τα οποία προβάλλουν στην αγορά. Θα δούμε τι θα γίνει λοιπόν. κύριο Σκυζίκα Κιζίκα, ευχαριστώ. Τέταρτη φορά και τελευταία. Να σας ρωτήσω το εξή. Οι προδιαγραφές για τις εκπομπές φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η τεχνολογία αυτή. Και σε ό,τι αφορά τα σωματίδια, θεωρώ ότι μπορούν να λυθεί το θέμα αυτό και τα σατούχα καλά πάνε. Ένα βασικό θέμα έχουμε με τα ντίζελ που είναι η ισορροπία σε ό,τι αφορά τα διοξείδια του άνθρακα. Το θέμα λοιπόν είναι τι θα προστατεύσουμε στην Αμερική, τι θέλει να προστατεύσετε την ε, υγεία του κάθε καταναλωτή ή το περιβαλλοντικό παράγοντα, το περιβάλλον. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αντίθεση. Πρέπει να σας πω ότι το diesel δεν βγήκε από την αγορά. Είναι δυνατή η πώληση, το, ε, η πώληση οχημάτων δίζελ στην αγορά. Ε, αυτή είναι μια επιλογή. Ε, το θέμα είναι να είναι καθαροί οι κινητήρες δίζελ και να κάνουν καθαρούς κινητήρες δίζελ ή ε, αυτοκινητοβιομηχανίες. Από την άλλη πλευρά, οι προσανατολισμοί της αγοράς ε, δεν μπορεί να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το πώς βλέπουμε εμείς ε, τον ντίζελ, κινητήρα. Θα είναι επιλογή της αγοράς και των αυτοκινητοβιομηχανιών. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσον θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη και τις επιλογές που θα κάνουμε, νομίζω ότι αυτές οι επιλογές είναι ε, Ε, θα πρέπει να κατασκευάζουμε ε, αυτοκίνητα τα οποία δεν θα εκπέμπουν οξύδια του αζότου ή διοξίδιο του άνθρακα. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον οι τεχνολογίες έτσι ώστε, ε, έτσι ώστε να δημιουργηθούν υβριδικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν την δυνατότητα χρήσης όλων των καλών τεχνολογιών και νομίζω ότι η αγορά μπορεί ωραιότατα να προχωρήσει κατά αυτή την έννοια. Σίγουρα δεν βγάζουμε εμεί οτιδήποτε από την αγορά, αλλά σίγουρα όλα, όλοι όσοι είναι παρόντες στην αγορά θα πρέπει να ε, δουλεύουν με το σωστό ανταγωνισμό. Μια ερώτηση. Γιατί είπατε ε, ότι είσαστε μηχανικός. Θα σας ρωτήσω λοιπόν σαν μηχανικός. Ε, μπορείτε να εξηγήσετε πως ένα αυτοκίνητο Ε, που ξεκινάει με ψυχρή εκκίνηση ε, μπορεί να έχει καλύτερη, ε, καλύτερη απόδοση από ότι ένα αυτοκίνητο που, που ξεκινά με θερμή. Αυτή ήταν τρίκη η ερώτηση, η απάντηση είναι όχι. Ναι, αλλά είπατε ότι 48 από τα 53 ελεγχόμενα αυτοκίνητα έδειξαν τέτοια συμπεριφορά. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω που το πάτε, είναι η απάντηση. Εγώ είπα απλά ότι και η ICCT και η Πολιτεία της Καλιφόρνιας όταν έκαναν ε, τις ε, ε, μελέτες probing questions as why this should be so. Ε, στα οχήματα της Volkswagen διαπίστωσαν αυτή την συμπεριφορά, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Άρα η απάντησή σας είναι ναι στην ουσία. Απάντηση. Πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω ε, γιατί ε, αυτά τα αυτοκίνητα έδειξαν μια τέτοια περίεργη συμπεριφορά. Εντάξει, ξέρατε είπατε που το πάω. Οπότε εγώ μπορώ να πω ότι αυτό ήταν... Ε, ε, ε, το η, ίδια η υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας απεκάλυψε ότι 48 από τα 53 αυτοκίνητα είχαν αυτή την συμπεριφορά αλλά σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε λέγοντας ότι ναι εσείς κάνατε την διαπίστωση αυτή ε, και επομένως ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί ε, υπόψη και από τη Volkswagen. Ναι. Μία τελική ερώτηση. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Διάβασα ότι είπατε στις γραπτές σας απαντήσεις ότι το σύστημα δεν είναι το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, στις ΗΠΑ δεν είναι απολύτως συγκρίσιμο, Αλλά και μετά από το σκάνδαλο της Volkswagen και στην Ευρώπη ε, βεβαίως έχει γίνει σαφές ότι χρειάζεται δοκιμασία αντί. και ε, στα μεμονωμένα κράτη-μέλη ε, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Ε, βεβαίως το επιχείρημα είναι ότι εάν προχωρήσει αυτό το αρντί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συσκευέ πλέον. Συμφωνείτε. Απάντηση. Θα είναι πιο δύσκολο. Εμείς κάνουμε διαφορετικές δοκιμές, μεταξύ των οποίων και η δοκιμή RD, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Αλλά προσπαθούμε μέσω αυτών να βρούμε κάποιες ε, περίεργες συμπεριφορές. Δεν αφορούν ακριβώς τη διαδικασία έγκρισης τύπου αυτή καθεαυτή. Βεβαίως ε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ε, τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι διαδικασίες RDE. Πρέπει πάντως να πω ότι το ΑΡΔΗ από μόνο του δεν είναι ικανοποιητικό. Θα πρέπει να προσθεθούν και άλλες διαδικασίες και άλλες ε, δοκιμασίες. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί, να αναπτυχθεί μια γενικότερη τεχνολογική ε, ικανότητα. Αυτή η τεχνολογική ικανότητα είναι απαραίτητη ε, έτσι ώστε να ε, υπάρξει πραγματικά να προωθηθεί η διαδικασία του καθαρού αέρα. Εάν θα ήθελα να, αν θα μπορούσα να κάνω, να δώσω μια συμβουλή που δεν θέλω γιατί είμαι ένας απλός μέσος Αμερικάνος, θα μπορούσα να πω ότι σαφώς έχετε μια τελείως διαφορετική κατάσταση με 28 ε, διαφορετικές ε, χώρες, αλλά θα τολμούσα να πω ότι δεν αρκεί κανείς ε, να έχει πολύ αυστηρά κριτήρια ή αυστηρές δοκιμές. Το ζήτημα είναι πώς εφαρμόζονται στην πράξη και πώς λειτουργούν σε σχέση με την ίδια την αγορά. Βεβαίως ε, ένα τέτοιο σύστημα επιβολής με 28 ξεχωριστές χώρες μέλη είναι σίγουρα ιδιαίτερα προκλητικό. Ε, Πρόεδρος, πρέπει να σας πω ότι για μας, ε, για το σύνολο της Επιτροπής μας αλλά και το σύνολο του Κοινοβουλίου, ο καθαρός αέρας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ Κοιτάξτε, εγώ αγαπώ την Ευρώπη, αγαπώ τους Ευρωπαίους πολίτες ε, και θα ήθελα να συνεχίσω και να ξαναέρθω και να εξεκολουθήσουμε να έχουμε επαφές. ευχαριστώ. If if there are some additional questions... Τώρα, εάν υπάρχουν επιπλέον ερωτήματα, μπορείτε να τα στείλετε μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου ε, στην Γραμματεία και εμείς θα τις προωθήσουμε ε, αρμοδίως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε.